Bueno, Λοιπόν, αν ε, συμφωνείτε, περνάμε στο σημείο 18 της ημερησίας διάταξης, παρουσίαση από το θεματικό τμήμα Β του ενημερωτικού σημειώματος με θέμα οι επιπτώσεις στην αλία εξατυχημάτων που αφορούν γεωτρήσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου και λαμβάνουν χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως ξέρετε, το θεματικό τμήμα ανέλαβε να συντάξει το ενημερωτικό αυτό σημείωμα και με τη σειρά του ανέθεσε τη σύνταξη του, θεματικού, του ενημερωτικού σημειώματος στο Πανεπιστήμιο του Αμπερντίν. Έχουμε λοιπόν το σημείωμα. Τι επίπτωση επίσης θα δούμε έχουν αυτά τα ατυχήματα στις ε, δραστηριότητες και θα ασχοληθούμε με τα πιο πρόσφατα ατυχήματα, τι αντίκτυπο έχουν θα δούμε και τι κόστος βέβαια πάνω από όλα αυτά και τι μέτρα μπορούν να υλοποιηθούν για την πρόληψη τέτοιων ατυχημάτων και για το μετριασμό των συνεπειών τους. Το ενημερωτικό σημείωμα λοιπόν είναι διαθέσιμο και έχει διανεμηθεί σε όλους δεν θα μακρηγορήσω, άλλο δίνω το λόγο στον συντάκτη του ενημερωτικού συμβιωματός, τον David Green, το Πανεπιστήμιο του Αμπερντίν, και τον παρακαλώ να μας παρουσιάσει. Έχετε 20 λεπτά, κύριε Green, στη διάθεσή σας για να μας κάνετε την παρουσίαση και μετά οι βουλευτές που ενδεχομένως το επιθυμούν θα ζητήσουν διευκρινήσεις ή μπορούν να έχουν μια ανταλλαγή απόψεων. Κύριε Green, καλώς ήρθατε στην Επιτροπή Αλίας, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την εισαγωγή σας. Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Λέγομαι David Green. Είμαι στο Πανεπιστήμιο του Αμπερτίν στο τμήμα γεωγραφίας. Η συνάδελφός μου η Κριστίνα Γκόμες δυστυχώς δεν μπόρεσε να έρθει μαζί μου σήμερα. Τι έρευνα κάναμε προσπαθήσαμε να δούμε ποιος είναι ο αντίκτυπος των γεωτρήσεων ε, για πετρέλαιο και για φυσικό αέριο ε, το, το αντίκτυπο των ατυχημάτων στις γεωτρήσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Αλία. This slide Εδώ βλέπουμε το περιεχόμενο της έρευνάς μας και συνάμα και τα κύρια αποτελέσματα αν θέλετε των ερευνών μας. Η έρευνά μας βασίστηκε σε βιβλιογραφική έρευνα πρώτα-πρώτα. Ε, ιστοσελίδες, δημόσιες ε, βάσεις δεδομένων. Είδαμε την νομοθεσία που επηρεάζει τις δραστηριότητες offshore στα ευρωπαϊκά είδατα και η σημασία των διαφόρων ατυχημάτων ε, τα χαρακτηριστικά τους, οι, τύποι των ατυχημάτων αναφέρονται εδώ και τέλος προσπαθήσαμε να, κάν, να έρθουμε και σε επαφή με φορείς που δουλεύουν στις γεωτρήσεις, παραδείγματος χάνει Shell, με την εταιρεία Shell. Λοιπόν, επειδή η Αλία είναι πολύ σημαντική για την Ευρώπη, εξετάσαμε και ε, μερικά πράγματα γενικώ για την αλία. Να δούμε ποιες είναι οι χώρες που αλλιεύουν, τι ποσοστά, ποια είναι η κοινή αλλιευτική πολιτική, ποια είναι τα αποθέματα των ισχυθείων ή τα είδη των ισχυθείων που ενδιαφέρουν και Βλέπουμε εδώ τώρα σε αυτή τη διαφάνεια την επικάλυψη των υδάτων ε, και εξόριξης πετρελαίου και φυσικού αερίου. Ιστορικά η περιοχή 2, δηλαδή τη Βόρεια Θάλασσα, περιοχή 2 και ήταν η μεγαλύτερη συγκέντρωση. Έκτοτε βέβαια έχουμε και στη Μεσόγειο επικάλυψη των υδάτων αυτών. Η κλάδη τώρα των, της εξόριξης πετρελαίου και φυσικού αερίου όπως επίσης και ο κλάδος ελίας, ακολουθούν συγκεκριμένους κανόνες Υπάρχουν και συμβουλευτικές επιτροπές στο Ηνωμένο Βασίλειο παραδείγματο χάρη η εταιρεία, μια εταιρεία του, που φτιάχτηκε το 2007 που ε, συνδέει αν θέλετε τους δύο κλάδους ε, πετρελαίου και αλίας Αυτές οι οργανισμοί κάνουν αρκετά καλή δουλειά. Εδώ βλέπετε τις οκτώ περιοχές που μας ενδιαφέρουν. Βλέπετε ποιες δραστηριότητες υπάρχουν εκεί και ποιο είναι το περιβάλλον μέσα στο οποίο γίνονται αυτές οι δραστηριότητες. Παράδειγμα, πάρτε την περιοχή 2, Βόρεια Θάλασσα. Εδώ πραγματικά οι εξορίξεις και οι γεωτρήσεις άρχισαν από πολύ παλιά. Άρα υπάρχει πείρα και πραγματογνωμοσύνη εδώ. Εμπειρογνω... και γνώση για την περιοχή και για τα νερά και για την πανίδα και για τη χλωρίδα και τα λοιπά. Η Shell ε, έχει κάνει λεπτομερή χαρτογράφηση στο, στις περιοχές αυτές ε, έχει φτιάξει iMaps ε, που είναι ουσιαστικά βάσεις δεδομένων για το περιβάλλον μα και στοιχεία που έχει πάρει από πάρα πολλά άλλα προγράμματα και έργα που έχουν γίνει. Για αυτή την περιοχή μιλάμε. Σε άλλες περιοχές όμως δεν, τα πράγματα δεν έχουν εξελιχθεί τόσο πολύ. Υπάρχουν βέβαια ιστορικά στοιχεία επί των οποίων μπορούμε να βασιστούμε και μπορούν να βασιστούν νέες δραστηριότητες. Παραδείγματο χάρη, ξέρουμε πολύ καλά ότι οι γεωτρήσεις είναι πιο δύσκολες σε πιο βαθιά ύδατα. Γιατί γιατί βεβαίω καινούργιες εξορίξεις πετρελαίου και φυσικού αερίου είναι σε μεγαλύτερο βάθος και εκεί πραγματικά οι γεωτρήσεις επηρεάζουν και πολύ περισσότερο τα αποθέματα εκθείων και την άρα και την αλία. Από όλες τις δραστηριότητες του ανθρώπου στο περιβάλλον ε, υπάρχουν συνέπειες για την πανίδα και τη χλωρίδα αλλά ειδικά για τις εξορίξεις πετρελαίου η διαρροή ε, πετρελαίου, οι πετρελαιοκυλίδες κτλ είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα που δημιουργεί τεράστια προβλήματα τα περισσότερα ατυχήματα που γίνονται στη θάλασσα και τα blowouts και οι εκρήξεις και τις μεταφορές και η κατάρρευση ε, κάποιες πλατφόρμας και τα χημικά δημιουργούν αυτές τις κοιλίδες και ε, οι κοιλίδες αυτές επηρεάζουν, ε, έχουν σημαντικές συνέπειες. Εδώ όλα εξαρτώνται από το μέγεθος της πετροκυλίδας, από τον τόπο που εμφανίζεται η κοιλίδα, από τον τρόπο μεταχεί, διαχείρισης της ε, κοιλίδας. Άμα πρόκειται για υδρατάνθρακες και κοιλίδα εκεί μπορούμε να ε, έχουμε τεράστιες συνέπειες ας πούμε στη, στο γόνο των ε, ψαριών. Επίση, οι πετρελοκυλίδες είναι πολύ πιο σημαντικές άμα είναι σε ριχά νερά ε, ή κοντά στην ακτή περιορισμένες κλειστές θάλασσες όπως τη Βαλτική, τον Άξινο Πόντο, τη Μεσόγειο είναι πιο σημαντικές οι συνέπειες γιατί δεν ανακυκλώνονται τα ύδατα εκεί πολύ συχνά όπως γίνεται στους ωκεανούς και στις ανοιχτές θάλασσες. Λοιπόν, ατυχήματα που γίνονται ε, τα ατυχήματα που γίνονται στη θάλασσα ε, καταγράφονται προφανώς και η βιομηχανία φυσικού αερίου και πετρελαίου είναι υποχρεωμένη να κοινοποιεί τα επεισόδια που συμβαίνουν ή τα ατυχήματα. Ιστορικά τώρα ε, μπορούμε να δούμε ότι η καταγραφή αυτών των ατυχημάτων ήταν αρκετά λεπτομερής και από πολύ παλιά μέχρι τώρα βλέπουμε ότι ε, καταγράφονται και, και τα ατυχήματα και οι κελίδες και τα λοιπά και αρκετές λεπτομέρειες γιατί, διότι παίρνουμε πάρα πολύ στα σοβαρά τα ατυχήματα και τις ε, διαρροές οι οποίες όπως σας είπα έχουν πολύ ε, κακές συνέπειες. Παράδειγμα, στο, στο διάγραμμα 3 του εδώ βλέπετε τα τι γίνεται με τα ατυχήματα τα τελευταία χρόνια. Βλέπουμε εδώ ότι πραγματικά όσον αφορά τον αριθμό των ατυχημάτων που γίνονται, ο αριθμός μειώνονται. Ε, γιατί, διότι τα τάνκερς, τα καινούργια τάνκερς είναι καλύτερα από τα παλιά, υπάρχει και, δηλαδή εδώ επεμβαίνει και τεχνολογία, ε, καινούργια τεχνολογία κτλ. Εδώ τα στοιχεία τα πήραμε από την παλιά UCOA, τώρα λέγεται OGUK, και βλέπουμε τον αριθμό των ατυχημάτων που γίνεται σε που έχουν συμβεί σε πλωτές μονάδες ή σε σταθερές μονάδες. Ε, μόντου, μόπου και μονού και λίφους. Στις πλωτές μονάδες τι γίνεται πέφτει ε, τα, ε, δεν έχουμε πολλές κοιλίδες ε, ΜΟΠΟΥ που είχαμε πολλές κοιλίδες και βλέπετε εδώ ότι τα περισσότερα ατυχήματα σχετίζονται με τις σταθερές μονάδες για, κατά την παραγωγή, όχι κατά τη γεώτρηση περιέργως. Επίσης όταν λέμε ατύχημα δεν σημαίνει ότι απαραίτητο το ατύχημα αυτό θα έχει ε, αντίκτυπο στην αλία. Ε. Again based on Λοιπόν και εδώ τα στοιχεία είναι από το OGUK την περίοδο 2000-2007. Βλέπετε ότι διάφορα ατυχήματα από τις διάφορες μονάδες γεωτρήσεων. Γεώτρηση μπορεί να γίνεται από διάφο, με διάφορους τρόπους, κινητές μονάδες, κινητές offshore ή κινητές ε, μονάδες παραγωγής και όχι γεωτρήσεων. Λοιπόν, εδώ βλέπετε, ε, εδώ βλέπετε τα ατυχήματα που συμβαίνουν, αλλά αυτά συνήθως δεν έχουν αντίκτυπο στην αλία. Αν κάνουμε μια ιστορική αναδρομή θα δούμε σε αυτό το πίνακα πως ότι η κύρια μόλυνση και οι περισσότερες κοιλίδες προέρχονται από τάνκερς, από μεταφορά φορτηγών, από πλοία φορτηγά που μεταφέρουν ε, διάφορες μορφές πετρελαίου, αργό ή όχι ή άλλο τα ατυχήματα είναι μοιραίο ότι θα συμβούν. Ό,τι και να κάνουμε για να ως πρόληψη είναι πολύ πιθανό να συμβούν ατυχήματα. Εδώ επηρεάζουν, ε, επηρεάζουν και καιρικέ συνθήκες. Παράδειγμα το Μπρέρ ε, το, και η σχετική κοιλίδα η οποία όμως διασπέζει διεσπάρει στη θάλασσα λόγω των ε, καιρικών συνθήκων επίσης. Α, πάντως η, σας λέω ότι εδώ μπορούν να γίνουν, ειδικά σε σχέση με τα σκάφη και τα τάνκερ μπορούν να γίνουν πολλά πράγματα με τις νέες τεχνολογίες. Ένα από τα 20 μεγάλα ατυχήματα των τελευταίων ετών έγινε στην Ευρώπη. Αυτά που βλέπετε εδώ, τα πρώτα, ε, αυτά που είναι σε κόκκινο είναι το Torrey Canyon, το Amoco Cadiz, Erin Serenade κτλ. Αυτά το έρικα Αυτά είναι τα πιο σημαντικά ατυχήματα τα οποία βέβαια προσήλκησαν και τεράστιο ενδιαφέρον της κοινή γνώμης. Ε. Ε, και στα οποία δόθηκε τεράστια δημοσιότητα. Το παλιό του 1967, εκείνη την εποχή ήμουνα στην Κορνουάλη εγώ, στο ατύχημα του Τόρι Κάνιον και ήταν πραγματικά πολύ ενδιαφέρον, ήμουνα καινούριο στα θέματα αυτά, να παρακολουθείς κανείς τι γινόταν. Τέλο πάντων... Βλέπετε εδώ στη φωτογραφία το σκάφος το οποίο τελικά έχει τραβηχτεί προς την ακτή, έχει σπάσει ή όχι και περιμένουμε να το καταστρέψουμε ουσιαστικά γιατί αυτό γίνεται συνήθως. Κάναμε λοιπόν την έρευνά μας και είδαμε τι άλλα, άλλες πηγές εκτός από το πετρέλαιο μπορούν να επηρεάσουν. Όπως για παράδειγμα θόρυβος, ε, ραδιενεργά υλικά, όλα αυτά αναφέρονται στη βιβλιογραφία και αυτά ε, δίνονται ως ε, περαιτέρω πληροφορίες. Επί τη βάση των όσων διαπιστώσαμε από το υλικό το οποίο συγκεντρώσαμε και διαβάσαμε, οι συγκεκριμένες αυτές πηγές ε, που θεωρούνται ως πηγές που έχουν συνέπειες δεν φαίνεται να έχουν ιδιαίτερες συνέπειες ε, για την αλληλεία και τα αποθέματα αλλιευμάτων. Ο θόρυβος για παράδειγμα μπορεί να οδηγήσει την ανακατανομή των ε, αλλιευμάτων και να επηρεάσει ίσως την γονιμοποίηση αλλά οι περιοχές τις οποίες τρέφονται τα αλλιεύματα και σε κάποιες περιπτώσεις ε, μπορεί να υπάρχουν ε, ζήματα σε ριχά νερά και να επηρεάσουν τα λιεύματα. Οι ατμοσφαιρικές εκπομπές ε, φαίνεται να μην έχουν καμία επιρροή στους πληθυσμούς των ελευμάτων και στην περίπτωση ραδιενεργού υλικού, από το υλικό το οποίο συγκεντρώσαμε, το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουμε είναι ότι οι ραδιενεργές εκπομπές από τις εξορίξεις και από τις πετρολοκυλίδες δεν φαίνεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει καμία συνέπεια ή μπορεί να μην υπάρξει συνέπεια σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά από τις ενδείξεις που έχουμε συγκεντρώσει, είναι μάλλον μικρή η επίδρασή του σε σχέση με τις άλλες δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα μια πετρελοκυλίδα. Να περάσουμε τώρα στον πυρήνα των ε, διαπιστώσεών μας. Υπάρχουν αρκετοί τρόποι με τους οποίους οι διάφορες δραστηριότητες εξόριξης, ε, όπως για παράδειγμα η ρήπανση που μπορεί να προκύψει από μια πετρελοκυλίδα, μπορεί να έχουν συνέπειες ε, στην αλία. Υπάρχουν άμεσες επιπτώσεις, μείωση της ζήτησης για παράδειγμα για την αλληλεία λόγω της άποψης της κοινή γνώμης, έμεσες επιπτώσεις ε, μέσω θνησιμότητας οργανισμών, ε, μείωση ε, στην παρουσία των ψαριών και αλλαγές στους ζωντανούς οργανισμούς και ε, έμεσες συνέπειες στα οικοσυστήματα. Οι περισσότερες από τις οποίες αυτή τη στιγμή δεν είναι και τόσο γνωστές, εξαρτώνται κυρίως από την δυνατότητα ανάπλασης του περιβάλλοντος και κάποιες συνέπειες δεν είναι και τόσο γνωστές. Δεν ξέρουμε για παράδειγμα και πολλά για τις μακροπρόθεσμες ε, συνέπειες των πετρολοκυλίδων στα ε, οικοσυστήματα, το κατά πόσο μπορεί να επιβιώσει το περιβάλλον και τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Ενδιάμεσες και μεσοπρόθεσμες ζημίες βέβαια στα οικοσυστήματα είναι πράγματα τα οποία μας ανησυχούν ιδιαίτερα, ιδιαίτερα αν η παραγωγή τροφίμων εξαρτάται από την ε, παραγωγή και καλλιέργεια ψαριών σε ηχθειοκαλλιέργειες κλπ. Επίσης μπορεί να επηρεάσουν και την αναπαραγωγική τους ε, δυνατότητα. Κάποιες από τις συνέπειες βέβαια είναι πιο προφανείς, ενώ κάποιες άλλες, ε, όπως σας είπα, ε, κάποιες υφέρπουν ή δεν είναι και τόσο γνωστές. Σύμφωνα με τις μελέτες ε, τις οποίες χρησιμοποιούμε σημείο αναφοράς, επειδή δεν ε, γνωρίζουμε κάποια πράγματα όσον αφορά τη δυνατότητα προσαρμογής των ε, ειδών και την στάση των αγορών, μπορούμε να μελετήσουμε αξιόπιστα μόνο τις βραχυπρόθεσμες συνέπειες. Όσον αφορά τώρα τις συνέπειες της αλληλείας ε, στις ε, ε, δραστηριότητες εξεόρυξης. Υπάρχουν ευρύτατα στοιχεία στη βιβλιογραφία. και ως προς τις άμεσες συνέπειες, ζημίας, εξοπλισμό, απολεχωρώνου εργασίας ή και έμεσες συνέπειες όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι μπορεί να ε, χαθεί η αξιοπιστία της κοινή γνώμης και η αποστροφή της αγοράς για κάποια είδη ε, αλλιευμάτων και να χαθούν έτσι και κάποιες ποσοστάσεις αντίληψη, το πώς αντιλαμβάνονται τις συνέπειες είναι ιδιαίτερα σημαντικές και σε περίπτωση των έμεσων συνεπειών ε, υπάρχουν και ουσιαστικές πτώσεις σε τιμές που μπορεί να ε, επηρεαστούν και από τη στάση των μέσων μαζικής ενημέρωσης και αυτό φυσικά επηρεάζει και τις τιμές και τις συνολικές ε, συνέπειες στην αγορά παρά το γεγονός ότι μακροπρόθεσμα η αγορά για ψάρια που αρχικώς είχαν χαθεί πολλές φορές ανακτούν τις τιμές τους και φτάνουν στα επίπεδα των προηγούμενων ε, τιμών πριν από κάποια, κάποιο περιστατικό. Ως παράδειγμα των όσων έχουμε διαπιστώσει για το οικονομικό κόστος ε, των συνεπειών που έχουμε, ε, πήραμε ένα παράδειγμα από μια μεγάλη καταστροφή. Το Πανεπιστήμιο του Αμπερντή συμμετείχε στην κατάρτιση μιας έκθεσης για την κυβέρνηση και εξετήσαμε τι έγινε στην καταστροφή αυτή μετά και η καταστροφή του Μπρέαρ, το οποίο βυθίστηκε πριν από κάποια χρόνια, είχαμε πολύ μεγάλες συνέπειες για τις αλληλευτικές δυνατότητες ε, και το 10% ε, των ε, were excluded for years των βενθόβιων λευμάτων ε, χάθηκε και όσον αφορά τα οστρακοειδή και αυτά είχαμε πολύ μεγάλες απώλειες. Υπήρχαν επίσης και συνέπειες για την αλληλεία που σε αυτή την περίπτωση αντιπροσωπεύουν ένα πάρα πολύ σημαντικό ε, ποσοστό απώλειας ε, και μάλιστα κυρίως σε μια συγκεκριμένη περιοχή, σε τοπικό επίπεδο δηλαδή. Από τις μεθόδους που αναπτύξαμε για την αξιολόγηση των οικονομικών συνεπειών υπάρχουν αρκετές μεθοδοί και δύο φαίνεται να προτιμώνται. Η μία είναι το κοινωνικό κόστος, το οποίο ορίζεται ως η αξιολόγηση της απώλειας εισοδήματος ε, ε, το διαφυγόν κέρδος δηλαδή ε, και πολλές φορές θεωρείται ότι αυτή είναι η οικονομική αξία της διαφοράς των εκφορτώσεων πριν και μετά το ατύχημα. Ε, χρησιμοποιήθηκε για παράδειγμα στην περίπτωση του πρεστή του Valdez και κάποια άλλα ως παράδειγμα. Η πιο απλή μέθοδος είναι η μέθοδος της αποζημίωσης το ποσό το οποίο δέχεται να πληρώσει ο αρμόδιος φορέας για την αποζημίωση θεωρείται ότι είναι το διαφυγόν κέρδος. Ε, ορισμένες φορές ε, ε, υπάρχουν κάποιες μέθοδοι οι οποίες μπορεί να είναι πολύ συγκεκριμένε, πολύ ακαδημαϊκές, πολλές φορές απαιτούνται δεδομένα τα οποία είτε δεν διαθέτουμε ε, σε νόμι, μόνιμη βάση ή δεν είναι πολύ εύκολο να τα βρούμε και πολλές άλλες μέθοδοι που δεν χρησιμοποιούνται περιλαμβάνουν και κάποιες μετολοποίησει. Και τα διδάγματα τα οποία αντλούμε είναι ότι οι μοντελοποιήσεις ε, δεν ε, είναι αποδεκτές γενικότερα από όλους όσους ε, δίνουν αποζημιώσεις, διότι δεν βασίζονται σε μεθόδους οι οποίες βοηθούν να γνωρίζουμε καλύτερα την αγορά. Ίσως γι' αυτό δεν την χάνουν και βρία συνένεση και ίσως θα πρέπει να υπάρχει και μεγαλύτερη υποστήριξη για να αναπτύξουμε κάποιες εναλλακτικέ μεθόδους, για να μπορέσει να υπάρχει μια βάση σύγκρισης όταν αξιολογούμε το οικονομικό κόστος και τις συνέπειες για την αλία. This slide, as an example illustration, summarizes the overall... Αυτό συνοψίζει τις συνολικές οικονομικές συνέπειες ε, με βάση τις ε, αγωγές για αποζημίωση. Υπάρχει ένα ταμείο αποζημιώσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο νομίζω ότι συστήθηκε το 1975. Και όπως βλέπετε, ε, ποικίλουν τα ποσά όσον αφορά τις αποζημιώσεις. Οι συνέπειες κυρίως αξιολογούνται από την απώλεια λευτικών εργαλείων ή η ζημία που γίνεται σε κάποιο σκάφος και δεν είναι πάντα σαφές αν όλα αυτά είχαν σχέση με πετρολοκυλίδες ή όχι. Κάποια από αυτά μπορεί να είχαν άμεση σχέση, αλλά μπορεί φυσικά να υπάρχουν και πολλοί άλλοι λόγοι για τους οποίους οι ελευτικές δραστηριότητες ε, μπορεί να μειώθηκαν. Μπορεί να μειώθηκαν γιατί υπήρξαν κάποια άλλα περιστατικά, τα οποία μπορεί να σχετίζονται βέβαια και με τις δραστηριότητες ε, της βιομηχανίας πετρελαίου και φυσικού αερίου. σοβαρά ε, ατυχήματα που περιλαμβάνουν πετρελοκυλίδες από πετρελαιοφόρα ε, μπορεί να έχουν πολύ μεγάλες συνέπειες σε σχέση με τον αριθμό των αλευμάτων που χάνονται. Ε, υπάρχουν ε, πολλά άλλες συνέπειες και όπως βλέπετε εδώ από τα στοιχεία τα οποία και πάλι ποικίλουν Έχουμε ως παράδειγμα για το οικονομικό κόστος ενός πολύ σοβαρού ατυχήματος, σε αυτή την περίπτωση του ατυχήματος του Πρεστή του 2002, το οποίο είχε συνέπειες για τις ακτές της Γαλλικίας και θα πρέπει εδώ να τονίσουμε ότι παρά το γεγονός ότι αυτός είναι ένας από τους τρόπους που μπορούμε να έχουμε αξιολόγηση του οικονομικού κόστους, η γενικότερη διεθνής βιβλιογραφία λέει ότι είναι δύσκολο να έχουμε αποτίμηση του πραγματικού κόστους γιατί λείπουν πολλά στοιχεία, ακόμα και τα στοιχεία των αλλιευμάτων που ε, δίνονται. Ε, υπάρχουν λοιπόν πολύ περίπλοκοι παράγοντες που δεν μας επιτρέπουν να βρούμε ε, ποιο ακριβώς είναι το οικονομικό κόστος για την αλληλεία και κάθε μέθοδος που εφαρμόζεται μας δίνει κάθε, κάποιο άλλο αποτέλεσμα. Και Ορισμένες φορές η αντίδραση για μια ε, τέτοια μορφή ατυχήματος μπορεί να οδηγήσει και σε διαφορετικές αλλευτικές δυνατότητες, μετατόπιση κάποιων περιοχών αλληλείας και μπορεί να υπάρχει και μικρότερη θνησιμότητα στην πραγματικότητα γιατί υπάρχει μια άμεση αντίδραση στην καταστροφή η οποία ε, είναι μια προσαρμογή την οποία σωστά πρέπει να λάβουμε υπόψη όταν αξιολογούμε το οικονομικό κόστος των συνεπειών. Παρά το γεγονό ότι το συγκεκριμένο ατύχημα δεν ήταν ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η περιβαλλοντική καταστροφή στον κόλπο του Μεξικού το 2010 από την Bison Horizon ε, ουσιαστικά επέστησε την προσοχή του κόσμου στο, ε, στις εξορίξεις αυτού του τύπου και τους κινδύνους και την ανάγκη να υπάρχουν κατάλληλοι κανονισμοί, αλλά επίσης αποτέλεσε και το ένευσμα για την ε, θέσπιση νέας νομοθεσίας η οποία στο μέλλον θα διασφαλίζει μεγαλύτερη ασφάλεια, τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Ε, αυτή τη στιγμή ε, ο βιομηχανικός ε, κλάδος πετρελαίου και φυσικού αερίου στα ευρωπαϊκά ύδατα έχει τις καλύτερες ε, προδιαγραφές ασφαλείας παγκοσμίως αλλά φυσικά ένα τύχημα μπορεί να συμβεί παρά τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνονται οι κίνδυνοι έχουν ελαχιστοποιηθεί με πολύ συγκεκριμένα μέτρα μετριασμού των συνεπειών, κατάλληλη πρόληψη, νομοθεσία και συγκεκριμένες συμβάσεις, ε, απόδοση ευθυνών και φυσικά έρευνα και τεχνολογία. Όσον αφορά την ε, συγκεκριμένη νομοθεσία και τις συμβάσεις, υπάρχουν πολύ περισσότερες λεπτομέρειες στην έκθεση, αλλά ως παράδειγμα θα μπορούσα να σας πω ότι για τη Μεσόγειο θα, Θάλασσα υπάρχει το πρωτόκολλο για τις εξορίξεις της Σύμβασης της Βαρκελόνης για την ε, Μεσόγειο Θάλασσα, υπάρχει Μαρπόλ, η Διεθνή Σύμβαση για την πρόληψη της ρήπανσης από τα αλλιευτικά σκάφη από τα σκάφη εν γέννη και υπάρχει και η σύμβαση της, του ευξήνου πόντου ε, κατά της ρήπανσης. Για την αποδόση ευθυνών υπάρχουν ε, για παράδειγμα κάποιες ενδείξεις από το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, η σύμβαση για την αστική ευθύνη για ζημίες από ε, ρήπανση από πετρέλαιο και στην περίπτωση της έρευνας και της τεχνολογίας νομίζω ότι είναι γνωστό ότι ο κλάδος του πετρελαίου και του φυσικού αερίου έχει πάρα πολύ ε, καλούς πόρους από χρηματοοικονομική σκοπιά και φυσικά επενδύει και σε έρευνα και ανάπτυξη τεχνολογίας, κάτι το οποίο φυσικά είναι θετικό. Υπάρχουν επίσης και μηχανισμοί για να μπορέσουμε να μετριάσουμε τις δυνητικές συνέπειες, όπως για παράδειγμα ε, την ανάγκη να υπάρχουν κάποια σχέδια δράσης, κάποια σχέδια εκτάκτου ανάγκης, ε, αποζημιώσεις και χρηματική αποζημίωση αλλά και πολλά μέτρα για να ε, βελτιώσουμε τα πράγματα για παράδειγμα η αφαίρεση των ρηπογόνων ουσιών ε, χημικές ουσίες που διαλύουν τις ε, διάφορες ε, ρηπογόνες ουσίες και φυσικά διεθνή συνεργασία και διεθνείς μηχανισμοί. Όσον αφορά τα ε, σχέδια εκτάκτου ανάγκης για τις πετρολοκυλίδες, έχουμε για παράδειγμα, δεν διαβάζω και τι γράφω εδώ, τη Διεθνή Σύμβαση για την ετοιμότητα για την ε, ρήπανση από πετρέλαιο, η οποία υπεγράφει το 1990. Όλα αυτά είναι διεξοδικότητα γραμμένα στην έκθεση, απλώς σας δίνω κάποια συνοπτικά παραδείγματα. Εδώ έχουμε κάποια παραδείγματα μηχανισμών τα οποία οι οποίοι δημιουργήθηκαν για να αντιμετωπίσουν τη σοβαρότητα των πιθανών συνεπειών όταν υπάρξει κάποιο σοβαρό ατύχημα για την Ευρωπαϊκή Αλληλεία. Στην ε, διαφάνεια 17, για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να έχουμε εδώ και το θέμα του Ταμείου Αποζημιώσεων των Αλλιέων. Όλα αυτά και πάλι, όπως σας είπα και προηγουμένως, προέκυψαν από την ανάπτυξη ενός ε, πλήρους ε, συνόλου εργαλείων για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε το περιβάλλον και στην έκθεση αυτή μελετούμε και τις δυνητικές συνέπειες από τις δραστηριότητες εξέριξης πετρελαίου και φυσικού αερίου. Ε, όλα αυτά καταδεικνύουν ότι υπάρχει ετοιμότητα η οποία ενισχύεται μέσω ελέγχου και κατάλληλων νομοθετικών μέσων που μας επιτρέπουν να μετριάσουμε τις συνέπειες, κατάλληλους μηχανισμούς για να μπορέσουμε να μειώσουμε τη ρήπανση και ε, να ελεγχεστοποιήσουμε τις πιθανές συνέπειες και τις οικονομικές και τις κοινωνικές και τις πολιτικές που μπορούμε να έχουμε σε συνέπεια ενός ατυχήματος. Ολοκληρώνοντας από πλευρά μου ατυχήματα συμβαίνουν, έχουν συμβεί στο παρελθόν και σε μεγάλο βαθμό, όπως διαπιστώσαμε μέσω αυτής της μελέτης, έχουν προκύψει ως αποτέλεσμα πετρελοκυλίδας, ε, το οποίο μεταφέρεται με πετρελοφόρα. Ε, και φυσικά αυτό συμβαίνει συνεχώς. Αλλά ο κόλπος του Μεξικού είναι ένα πολύ καλό και πρόσφατο παράδειγμα του τι μπορεί να συμβεί παρά τις ε, τα μέτρα τα οποία μπορεί να έχουν θεσπιστεί και όλα τα μέτρα ασφαλείας τα οποία μπορεί να έχουν ληφθεί. Ο κλάδος του πετρελαίου και του φυσικού αερίου έχει εκτεταμένη γνώση, χρήματα και ε, αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει, κυρίως από τις δραστηριότητες στη Βάρια Θάλασσα από τη δεκαετία του 70 και αυτό μας ε, βοήθησε να υπάρχει μια καλή βάση για τις δραστηριότητες εξαίρεσης πετρελαίου και φυσικού αερίου. Υπάρχουν κατάλληλα μέτρα για αποζημιώσεις και υπάρχουν και επειδή υπάρχουν δυνατότητες να υπάρχουν εξορίξεις και σε άλλες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της οδηγίας 2013-30, Ευρωπαϊκή Νομοθεσία την οποία φαντάζομαι ότι γνωρίζετε, επικεντρωνόμαστε στην ασφάλεια των παράκτιων εξορίξεων καθορίζονται κανόνες για όλο τον κύκλο ζωής ε, πετρελαίου και φυσικού αερίου, και ε, ανταλλαγή πληροφοριών, ε, ε, υπεύθυνη αντίδραση και το καθεξής. Πολλά πράγματα περιλαμβάνονται στην οδηγία. Τέλος, έχουμε κάποιες συνοπτικές συστάσεις σε διάφορες θεματικές ενότητες. Όσον αφορά στα ρυθμιστικά μέτρα, θέλουμε να επικεντρωθούμε στην οδηγία 2013-30, να μεταφερθεί αυτή στο εθνικό δίκαιο, ώστε να διασφαλίσουμε ότι υπάρχουν κατάλληλοι μηχανισμοί εφαρμογής, υπάρχει ανάγκη ρυθμιστικών πλαισίων και φυσικά να τηρούνται οι κανόνες και να διασφαλίζεται ότι όλα αυτά θα γίνονται ασφαλώς όσον αφορά το διεθνές περιβάλλον θα πρέπει να υποστηρίξουμε αυτή την αναδυόμενη βιομηχανία και εδώ ίσως θα έπρεπε επειδή υπάρχουν και νέες εξοριστικές ε, δραστηριότητες οι οποίες ήδη έχουν ξεκινήσει σε κάποια ε, ευρωπαϊκά ύδατα και θα αποτελέσουν πρόκληση για τον κλάδο του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, διότι θα υπάρχουν νέες περιβαλλοντικές συνθήκες και θα πρέπει φυσικά να εφαρμόσουν και όλα τα διδάγματα τα οποία έχουν μάθει στο παρελθόν και φυσικά υπάρχουν και πολλά διεθνή παραδείγματα για το τι θα μπορούσε να συμβεί. Επιπλέον, για να προωθήσουμε προδιαγραφές ασφαλείας και κανονισμούς στις γειτονικές χώρες, θα πρέπει να δοθεί κάποια έμφαση και σε αυτό. Όσον αφορά την έρευνα και την τεχνολογία, θα πρέπει να προωθήσουμε την έρευνα και την ανάπτυξη σε συγκεκριμένε δραστηριότητε, εξορυκτικές δραστηριότητε και να διασφαλίσουμε φυσικά ότι θα υπάρχει συνεχής χρηματοδότηση για όλες τις πηγές και όσον αφορά τις αποζημιώσεις τώρα να προσπαθήσουμε να βελτιώνουμε τις μεθόδους αξιολόγησης για το οικονομικό κόστος, ε, δεδομένα τα οποία απαιτούνται για να μπορέσουμε να αποζημιώνουμε για ε, ατυχήματα και να υπάρχει αποζημίωση για όλους τους σχετικούς τομείς, να προσπαθήσουμε να καλύψουμε ακόμα και κάποιες συνέπειες τις οποίες δεν αντιλαμβανόμαστε επαρκώς όσον αφορά τη χωρική και χρονική διάσταση. Να σας ευχαριστήσω λοιπόν για την προσοχή σας, για το χρόνο που με διαθέσατε και για το γεγονός ότι μας δώσατε την ευκαιρία να κάνουμε αυτή την έρευνα και τέλος να ευχαριστήσω τον Ραφαέλ για τη συνεχή του υποστήριξη και γιατί ε, υπέστη όλων αυτό των οριμαθό των ερωτήσεων για πάρα πολύ καιρό. Ευχαριστώ πολύ. Muy bien, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Γκριν για την ενδιαφέρουσα αυτή παρέμβαση. Θα ξεκινήσει ο συνήθως ένας γύρος ε, ρωταπαντήσεων Λοβίν και Ρόντουστ. Κυρία Λοβίν, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Γκριν, ε, σας ευχαριστώ πολύ για την ε, πληρέστατη αυτή διεξοδική παρουσίαση. Αν κατάλαβα, Πολλοί είναι οι παράγοντες που δεν ξέρουμε και πολύ καλά πόσο μπορούν να περάσουν το περιβάλλον και ιδίως τα ηχθή αποθέματα. Κάτι που αναφέρατε στο τουλογική έκθεση είναι ότι τα μικρής κλίμακας ατυχήματα, μικρές πετρελοκυλίδες που φαντάζομαι ότι είναι καθημερινή υπόθεση χωρίς να γίνεται πρωτοσέλιδο. Θα ήθελα να μας πείτε λίγο πιο αναλυτικά τι αντίκτυπο θα μπορούσαν να έχουν αυτές οι μικρές πετρελοκυλίδες στο περιβάλλον και συγκεκριμένα στα τα αποθέματα. Και σε ό,τι αφορά το κόστος, φυσικά και υπάρχει δυνατότητα να μετρήσει κανείς το κόστος, την αντιστάθμιση, την αποζημίωση που δίνεται δηλαδή στους ψαράτες και έτσι να προσπαθήσει να υπολογίσει το κόστος των ατυχημάτων των πετρελοκυλίδων που δημιουργούνται. Ίσως να υπάρχουν και άλλοι τρόποι βέβαια για τον υπολογισμό του συνολικού αντικτύπου αυτών των περιβαλλοντικών ατυχημάτων στο οικοσύστημα. Αυτό φαντάζομαι ότι είναι πιο δύσκολο να υπολογιστεί δηλαδή αντίκτυπος στον τουρισμό ή στα από θέματα μακροπρόθεσμα. Δεν ξέρω μήπως δεν πρόσεξα, αλλά αναφέρατε μήπως ε, τα συνολικά ποσά αποζημίωσης που πηγαίνουν σε Ευρωπαίους αλείς ή αλείς στην Ευρώπη. Λόγω ατυχημάτων ε, με πετρελαφυσικό αέριο. Αυτές είναι οι ερωτήσεις μου, Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Να δώσω πρώτα το λόγο στον κύριο Ρόντουστ και θα απαντήσει εν συνεχεία και στις δύο σας ο κύριος Γκριν. Μπορείτε να απαντήσετε μετά κύριε Γκριν. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Γκριν, και εμένα μου άρεσε πολύ η παρουσίασή σας. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Σας ευχαριστώ για την παρουσίαση αυτή. Αλλά έχω δύο ερωτήματα να σας θέσω. Πιστεύετε μετά από την έρευνα που κάνατε ότι το πρόβλημα το παίρνουν στα σοβαρά όλοι οι ενδιαφερόμενοι διότι ε, τα, τάνκερ και τεχνολογία διπλού και λύφους για τάνκερ ας πούμε παρά, που κοστίζουν παραπάνω βεβαίως και ε, δεν ξέρω αν θυμάστε στη Βαλτική ένα τύχημα που έγινε τότε η σαν σύσταση ε, είχε λεχθεί ότι πρέπει να είναι διπλού και λίφους τα τάνκερ τα οποία κοστίζουν περισσότερο βεβαίως και σε τελευταία ανάλυση Άμα γίνει το ατύχημα, ποιος πληρώνει αυτός που δημιούργησε το ατύχημα ή ο φορολογούμενος. Μικρές κοιλίδες, ναι, δημιουργούν μικρέ, έχουν μικρές συνέπειες, αλλά τελικά μακροπρόθεσμα θα ε, υπάρξει κάποια ζημιά στο περιβάλλον. Ποιος θα το πληρώσει αυτό, ο φορολογούμενος ή ο αυτός που ήταν που δημιούργησε τις κοιλίδες αυτές. Εμείς σαν ευρωβουλευτές τι μπορούμε να κάνουμε. Έχω την εντύπωση ότι τώρα, με, ιδιαίτερα μετά και τη δική σας έρευνα, ξέρουμε πάρα πολλά πράγματα. Αλλά δεν ε, ξέρουμε τι να κάνουμε. Ε. Ο κύριος Γκριν να απαντήσει. Ευχαριστώ πολύ, αλλά ε, χωρίς μικρόφωνο. Μ' ακούτε τώρα? Μάλιστα. Κάτσω και πιο κοντά. Νομίζω ότι αναφέρατε αρχικά τα μικρότερη κλίμακα ατυχήματα. Φαντάζομαι ότι γενικά πολλά από αυτά δεν γίνονται τόσο γνωστά οι περισσότερε γνώσει ε, που αποκομίσαμε είχαν να κάνουν με μεγάλες κλίμακες ατυχήματα τα οποία βοηθούντων και των μέσων ενημέρωση πήραν μεγάλη δημοσιότητα. Φυσικά υπάρχουν και μικρές κλίμακες ατυχήματα. Τώρα κατά πόσον αυτά θεωρούνται ότι έχουν κάποιο αντίκτυπο στην αλία επειδή είναι πολύ ε, τοπικά, εντοπίζονται σε μικρό διάστημα, ε, μάλλον δεν έχουν ή δεν υποτίθεται ότι έχουν πολύ μεγάλο αντίκτυπο. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να τα δούμε από πλευρά επιστημονικών μελετών του Σύνηγκης. Επίσης, διαβάσαμε τη βιβλιογραφία και είναι μελέτες πολλές που είναι περιορισμένες σε ένα συγκεκριμένο τοπικό, ε, σε μια μικρή περιοχή. Οπότε, φαντάζομαι ότι υπάρχει ανάγκη να μελετήσουμε και αυτά τα μικρά ατυχήματα συμβάντα για να είμαστε βέβαιοι ότι δεν έχουν ένα σημαντικό αντίκτυπο και αυτά. Για παράδειγμα, ίσως έχει γίνει ε, κάποιο σχετικό έργο, αλλά δεν βρήκαμε κάτι γι' αυτό. Δεν βρήκαμε δηλαδή στη βιβλιογραφική μας αναζήτηση κάτι. Τώρα, αν δει κανεί τη ρήπανση από βαρέα μέταλλα, για παράδειγμα, ιστορικά, σε, μακρι... σε μεγάλη κλίμακα ε, δεν φαίνεται να έχουν μεγάλο αντίκτυπο, αλλά αν αρχίσει κανείς να ψάχνει, βρίσκει μικρά ποσοστά ε, ρήπανσης που όμως τελικά τελικά επηρεάζουν πολύ περισσότερο το σύστημα από όσο νομίζαμε στην αρχή. Και αυτό ίσω να συμβαίνει και με τι πετρελοκυλίδες. Δεν μπορώ όμω να σα δώσω ε, μια πιο λεπτομεριακή απάντηση. Είναι σίγουρα ένα τομέα που πρέπει να ερευνηθεί και πιστεύω ότι θα πρέπει να διεξαχθούν περισσότερες επιστημονικέ μελέτε που να μην εστιάζουν τόσο σε συγκεκριμένα πράγματα, αλλά γενικότερα στον αντίκτυπο των ε, δραστηριοτήτων ε, γεώτρηση και πετρελαίου και εξόρυξης φυσικού αερίου. Πάντως δεν βρήκαμε και πολλά στοιχεία. Ε, δεν βρήκαμε κάποιες γενικές ε, μελέτες πιο συγκεκριμένες. Τώρα κάτι που πράγματι ε, ξέχασα. Α, ναι, ήταν αυτό το κόστος μάλιστα. Βρήκαμε κάποια παραδείγματα. Τις μεθόδους τις μελετήσαν. Πολλές από αυτές ήταν ακαδημαϊκές εστίασαμε σε κάποιες από αυτές δεν ήταν πιο ρεαλιστικές ούτε οι πλέον κατανοητές ό,τι αφορά το πώς ε, ε, προέκυψε η αποζημίωση και πού δόθηκε, τι δόθηκε ως αποζημίωση κτλ. Στο τέλος των συστάσεων όμως, ναι, πράγματι λέω ότι υπάρχει η ανάγκη να δούμε πιο προσεκτικά τους μηχανισμούς αντιστάθμισης αποζημίωσης και να μελετήσουμε και άλλες μεθόδους. Γιατί κάποια από τα παραδείγματα που δεν σας τα ανέφερα σε αυτήν την παρουσίαση, πράγματι ε, μας κάνουν να πιστέψουμε ότι υπάρχουν ε, διαφορές. Με τη μέθοδο αλλάζει και το αποτέλεσμα και είναι δύσκολο να φτάσουμε σε μία απάντηση ε, που να είναι και τελεσίδητη κατά κάποιο τρόπο. Αν δει κανείς τις μεθόδων, αυτών των μεθόδων, ε, προφανώς υπάρχει κάποια ανησυχία. Μήπως κάποιες από τις απλές μεθόδους ίσως παρά είναι απλές τελικά. Ναι, μεν βοηθάνε γιατί εύκολα μπορεί κανείς ε, να διαβάσει τα αποτέλεσμα των μεθόδων αυτών, αλλά καλό θα ήταν ίσως να μελετήσουμε άλλες μεθοδολογίες και πώς συγκρίνουμε ε, ε, την μικρή κλίμακα με την ευρύτερη κλίμακα. Μάλλον δεν έχει γίνει ακόμη πολύ στο κομμάτι αυτό. Άρα καλό θα ήταν να μελετήσουμε τις μεθόδους για να μπορέσουμε να δώσουμε μια πληρέστερη απάντηση. Δεν ξέρω αν σας βοηθά αυτή η απάντηση. Κάπως, μάλιστα, ωραία τώρα. Πρέπει να απαντήσω και τα δικά σας ερωτήματα. Δεν θα έπρεπε μάλλον τα είχα γράψει γιατί δεν θυμάμαι τίποτα, τέλος πάντων. Δεν μου θυμίζετε, σας παρακαλώ. Ποιο ήταν το πρώτο σας ερώτημα. Γρήγορα έτσι να τα πω περιεκτικά. Μίλησα ουσιαστικά για το ποιος πληρώνει. Πληρώνει αυτός τον ο οποίος δημιουργεί το ατύχημα ή πληρώνει ο φερολογούμενος. Έχετε την εντύπωση ότι αναγνωρίζουν οι πολιτικοί το πρόβλημα ε, ή απλώς θέλουν να τελειώνουν με την όλη ιστορία και ζητούν ας πούμε από τους φορολογούμενους ή προσπαθούν μέσω των, των χρημάτων των φορολογουμένων να αποζημιώσουν όσο πιο γρήγορα γίνεται χωρίς να ε, ψάξουν για το ποιος έφταιγε κτλ. Δηλαδή πιστεύετε ότι η πολιτική έχει συνειδητοποιήσει τη σοβαρότητα του θέματος. Okay, thank you very much. Okay. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ. Για κάποια από τα παραδείγματα που μελετήσαμε, περιλαμβάνονται στην ε, έκθεση, όχι όλα φυσικά, και σίγουρα επικεντρώνονται σε αυτή την αρχή ορυπαίνων πληρών. Όχι ο φορολογούμενος. Δεν θέλω να σχολιάσω τι πληρώνει ο φορολογούμενος βέβαια, γιατί δεν μελέτησα αυτή την πτυχή. Εμείς Είδαμε αυτή την αρχή ε, και βλέπουμε ότι ο Ριπένων είναι αυτός ο οποίος πρέπει να λάβει την ευθύνη και να πληρώσει. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη δεύτερη ερώτησή σας, υποπτεύομαι ότι η ευαισθητοποίηση της κοινή γνώμης δεν είναι και τόσο μεγάλη. Νομίζω ότι πολλέ φορέ τα μέσα μας και ενημέρωση παραφουσκώνουν, διωγγώνουν τα πράγματα. Κάποιε φορέ όμω έχουν και ένα θετικό ρόλο γιατί στρέφουν την προσοχή του κόσμου τη κοινή γνώμη σε κάποια τέτοια ατυχήματα. Ο αντίκτυπος ε, είναι σημαντικό για έναν άνθρωπο αν γίνει στην περιοχή που μένει, υποθέτω. Εκεί δηλαδή που είναι και ορατό ο αντίκτυπο ε, και γίνεται αισθητό. Αλλού, τώρα σε ό,τι τα δεξαμενόπλια ε, πετρελαίου, υπήρξαν αλλαγέ στην τεχνολογία, μιλήσατε για το διπλό κέλυφος, διπλό κήτος. Έχει ελαχιστοποιηθεί. Ο κίνδυνο δεν έχει αποτραπεί εντελώ βέβαια, ε, ο κίνδυνο πετρελοκυλίδα. αλλά σίγουρα η όγκη, ε, ο όγκος ε, πετρελοκυλίδων έχει μειωθεί. Και η μεταφορά που γίνεται με τα πλοία έχει μειωθεί. Άρα μειώνονται και τα ατυχήματα. Σίγουρα έχουμε να διδαχθούμε πάρα πολλά σε ό,τι αφορά ε, τις δοκιμαστικές γεωτρήσεις, ε, πετρέλαιο φυσικό αερίου σε άλλες περιοχές, σε νέες περιοχές. Και αυτό πρέπει να το ε, μελετήσουμε πολύ περισσότερο από ό,τι μέχρι τώρα. Πάντως γνώση υπάρχει. Ε, νομίζω υπάρχει ευαισθητοποίηση, δεν ξέρω αν φτάνει στα σωστά άτομα, εκεί που πρέπει, αλλά πιστεύω ότι μεγάλο μέρος των πληροφοριών που σταδιακά γίνονται πιο διαφανείς και δημοσιοποιούνται έτσι πιο ελεύθερα, επιτρελακές εταιρείες υποτίθεται ότι γίνονται πιο φιλοπεριβαλλοντικές και πιο πράσινες, ίσως όχι βέβαια γιατί θέλουν να σταματήσουν τη ρήπα κατά ανάγκη, αλλά τέλος πάντων. Πάντως υπάρχει μια μετατόπιση σταδιακή προς ε, την ε, απόδοση μεγαλύτερης σημασίας ε, στον πολύ σημαντικό αυτό ε, ορυκτό πλούτο και για την προστασία του παράκτου περιβάλλοντος, αλλά έχουμε ακόμη δρόμο να διανύσουμε για να ενημερώσουμε τον κόσμο και να δώσουμε μια σωστή εικόνα για το πώς λειτουργούν οι εταιρείε πετρελαίου φυσικού αερίου, πόσο υπεύθυνα συμπεριφέρονται, τι κάνουν σε περίπτωση διαρροών, απορρίψεων πετρελαίου ή τι κάνουν σε περίπτωση καταστροφών όπως αυτή στον κόλπο του Μεξικού σε κάποια κομμάτια, σε κάποια μέρη μάλλον του κόσμου, είναι σαφές ότι παρά τις προσπάθειες ή τις υποτιθέμενες προσπάθειες, δεν αρκούν αυτές πάντοτε. Και αυτή η τις υποτιθεμενες προσπαθειες δεν αρκουν αυτες παντοτε και αυτη η παναξιολογηση του αντίκτυπου αυτών των δραστηριοτήτων για ότρες πίεσης πετρελαίου φυσικού αερίου νομίζω ότι είναι κάτι πάρα πολύ επίκαιρο. Είναι σωστό το timing και πολύ σημαντικό βέβαια το timing. Υπάρχουν πολλές άλλες προκλήσεις, πολλά γίνονται στον τομέα αυτό και η τεχνολογία προσπαθεί να υπερκεράσει κάποια από τα εφιστάμενα προβλήματα και η νομοθεσία φυσικά γίνεται πιο αυστηρή. Αλλά πιστεύω ότι ξεκολουθούν πολλά να πρέπει να γίνουν και στον τομέα των επιστημονικών μελετών. Πρέπει να μελετηθεί περισσότερο αντίκτυπος των δραστηριοτήτων γεωτρήσεων ή πετρελοκυλίδες, ε, τα blowouts ε, αναρροέ κτλ. Όλα αυτά δεν τα γνωρίζουμε πολύ καλά, δεν γνωρίζουμε ποιε είναι οι μακροπρόθεσμε επιπτώσει. Για το εξονβαλτές, για παράδειγμα. Ήταν θετικέ εξέλιξει με την έννοια ότι ε, επιδιορθώθηκε πιο γρήγορα η κατάσταση. Αλλά στον Μπρέαρ, για παράδειγμα, ο αντίκτυπο ε, διήρκεσε για δύο χρόνια. Η επιπτώση των ορατέ δύο χρόνια. Κατά τύχη όμως επειδή ευνόησαν και οι καιρικέ συνθήκες εκείνο τον καιρό, δεν έγιναν πολύ χειρότερα τα πράγματα. Αλλά σίγουρα πρέπει κανείς να βλέπει πώς επηρεάζει ο καιρό, ο χρόνος, ποια είναι η κλίμακα, αν έγινε σε τοπικό επίπεδο, πιο ευρύ, και τελικά να δούμε αν το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο μπορεί να επηρεάσει και να έχει έναν αντίκτυπο πιο μακροπρόθεσμο και σε μια ευρύτερη περιοχή, πέραν τη στενή γεωγραφική περιοχή που έγινε το ατύχημα. Πρόεδρε, σα ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν ερωτήσει άλλε. Όχι. Άρα ε, να ευχαριστήσουμε τον κύριο Γκριν και να τον αποχαιρετήσουμε. Περνάμε στο σημείο 19 της μερικής διάταξης. Διάφορα. Εγώ θεωρώ ότι τα έχουμε καλύψει όλα. Υπάρχει κάποιο θέμα που θέλετε να θέσετε, όχι. Οι βουλευτίνες που έμεναν εδώ δεν έχουν να θέσουν κάποιο θέμα, άρα πάμε στην προσεχή συνεδρίαση. 10 Φεβρουαρίου, μάλλον 11 Φεβρουαρίου ο πρόεδρος, το πρωί και το απόγευμα. Σας ευχαριστώ όλους και τους διερμηνείς και κύριε τη της συνεδρίας.